Ε. Πασκάλ δεν είναι εδώ. Άλλος κανείς δεν ζητεί το λόγο από ό,τι φαίνεται. Άρα λοιπόν εσείς Σοφή. Δεν ε, λύθηκαν τα προβλήματά μου κυρία Πρόεδρε. Σημειώνω τις σκέψεις που εξέφρασε ο Πίτερ. Ε, είμαι διαθέσιμη για οποιαδήποτε συζήτηση με ενδιαφερομένους συναδέλφους όταν θα έχουν εξετάσει ολόκληρο το φάκελο για να με βοηθήσουν ε, στην περαιτέρω εργασία για να κλείσει ο φάκελος. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 15 Τρίτου. Υπάρχει λοιπόν ακόμη χρόνος για τις σχετικές συζητήσεις. Η ψηφοφορία στην αρμόδια ψηφιακή επιτροπή θα γίνει τον Απρίλιο και στην Ολομέλεια τον Ιούνιο. Ας προχωρήσουμε λοιπόν τώρα στο θέμα υπαριθμών 4 της ημερήσιας διάταξης που αναφέρεται στην τροποποίηση του άρθρου 136 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς θα χρειαστεί να φύγω ακριβώς στις 11 ή και λίγο πριν δεν φεύγω διότι θεωρώ ότι δεν είναι σημαντικό ε, το θέμα, αλλά ίσως προλάβουμε να ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις μας μέχρι εκείνη την ώρα. Ε, είστε εδώ, Έντουαρτ. Α, ναι, ναι. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η αίθουσα γιατί δεν βλέπω τους συναδέλφους μου καλά. Έντουαρτ, λοιπόν. Θα ήθελα καταρχήν να σας πω ότι συζητούμε εδώ τη συμπερίληψη ενός άρθρου στην συνθήκη που δεν προϋπήρχε. Και δεν προϋπήρχε διότι τότε είχε θεωρηθεί ότι ο αποκλεισμός αυτού του άρθρου θα είχε οδηγήσει την ανάσχεση της χρηματοπιστωτικής κρίσης σε επίπεδο κρατών μελών. Είδαμε ότι αυτό δεν μάλλον η κρίση συνέβη. Και γι' αυτό αυτός ο μηχανισμός θα πρέπει να προβλεφθεί. Τουλάχιστον αυτά είναι τα σχόλια που έχουμε λάβει, δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα σχετικός μηχανισμός, αλλά δεν συμφωνούμε ως προς το τι θα περιλάβει και τι θα πρέπει να συμπληρώσει αυτό το μηχανισμό. Βεβαίως πολλέ, πολλά ζητήματα αρχής αναφέρουν, δηλαδή το θέμα των ε, ισολογισμών, των ανισορροπιών ή την, των διαφορών μεταξύ κρατών μελών ως προς θέματα αντιστάθμισης. Δεν ξέρουμε πώς να τα αντιμετωπίσουμε και γι' αυτό ε, προβλέφθηκε και το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης. Θα πρότεινα λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί και στην έκθεσή μας να μην θέσουμε λεπτομέρειες και να προβλέψουμε ειδικά μέτρα αντιστάθμισης, τα οποία δεν έχουν συζητηθεί εκτενώς, εκεί δηλαδή όπου δεν υπάρχει απόλυτη συνένεση. Επίσης όμως δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε Δεν πρέπει να αποκλείσουμε δυνατότητες και συμπληρωματικά μέτρα αντιστάθμισης στο μέλλον. Το τελικό θέμα αφορά τη διατύπωση. Είδα πολλές ε, τροπολογίες, είδα τις τροπολογίες, υπάρχει συμφωνία. Αν λοιπόν είμαι βέβαια αισιόδοξο, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε συνένεση. Υπάρχει όμως μία τάση που διαγράφεται, που δείχνει ότι η διατύπωση του Συμβουλίου είναι κάπως περιοριστική και όχι απόλυτα ε, σαφής όταν μιλάμε για τη σταθερότητα του ευρώ, όταν μιλάμε για τα μέλη της Ευρωζώνης. Μέλη της Ευρωζώνης που συνεισφέρουν σε αυτόν τον κανονισμό, τους ε, καθαρούς εισφορείς δηλαδή, και εκείνους που θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρχει μία αρχή επικουρικότητας, ελπίζοντας ότι εάν χρειαστούν ένα παρόμοιο μηχανισμό δεν θα υπάρχει κανένα ερωτηματικό. Δηλαδή σίγουρα θα λάβουν αυτή την ε, ενίσχυση. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να το κάνουμε αυτό, αλλά θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα μέλη της Ευρωζώνης είναι μια οικογένεια. Θα πρέπει να υπάρχει ένα στοιχείο αλληλεγγύης. Όλοι έχουν, όλοι συνεισφέρουν, άρα δεν θα πρέπει να αποκλειστούν. Για, ως προς την αρρωγή που υπάρχει, που υπάρχει και θα πρέπει να αντιλάβουν αν είναι αναγκαίο. <coughs> Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον συνεισηγητή. Συμμεριζόμαστε την προσέγγιση αυτή. Χτες συμμετείχα σε ένα συμπόσιο για την συνθήκη της Λισαβόνας και είχαμε έναν ε, ε, καθηγητή δικαίου από τη Γερμανία που εκπροσωπεί το ε, Bundestag ενώπιον του συνταγματικού δικαστηρίου της Καρλσρούης. Δυστυχώς δεν ήταν καθόλου καθησυχαστικά αυτά που μας είπε, διότι το γεγονός ότι εισαγάγουμε αυτό το νέο ε, άρθρο στη συνθήκη, το σημείο Γ, δεν εγγυάται ότι θα υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Και δεν θα ε, βρεθούμε ενώπιον μιας διαδικασίας αντιμετώπισης. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε ποια είναι η προσέγγιση που ε, προβάλλουμε και κατά πόσο προτρέχουμε. Το δεύτερο ζήτημα στο οποίο γνωμοδοτούμε είχε υποβληθεί από το Συμβούλιο και θα πρέπει να είμαστε σίγουροι για το πώς θα τροποποιήσουμε αυτό το κείμενο. Νομίζω, όπως είπε και ο συνεισήγητης, ότι με βάση αυτή την έκθεση μπορούμε να υποβάλουμε υποδείξεις, ιδέες στην αιτιολογική σκέψη έτσι ώστε να υπάρχει ευρία αλληλεγγύη ως προς την Ευρωζώνη αλλά ως προς το κείμενο δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Όμως με βάση τη γνωμοδότηση του Μέντες Δεβίγκο και μαζί με τον Έντουαρντ Σικλούνα μπορούμε στην τροπολογία 23 να δούμε πώς μπορούμε να προβάλλουμε αυτό τον συμβιβασμό η οποία θα αντικαταστήσει την αρχική σε σχέση με την τροποποίηση του 3Γ. Νομίζω ότι αυτό το κείμενο βρίσκεται στα πλαίσια αυτού που πραγματικά μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή να λάβουμε υπόψη ορισμένα στοιχεία που έδωσαν και η ΜΕΝ και η ΔΕ. Γι' αυτό επιμένω σε αυτή την πρόταση 23 που είναι μια κοινή πρόταση που θα δείτε ότι αναφέρεται σε πολλά στοιχεία των τροπολογιών που υπέβαλαν οι μεν και οι δε, έτσι ώστε αυτό το κείμενο να είναι συνεκτικό και συνεπές με αυτό που προτείνουμε στο Κοινοβούλιο γενικότερα. Αυτά σε σχέση και με αυτά που προείπε ο άλλος εισηγητής. Θα δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε στο κείμενο. Ορισμένες τροπολογίες ε, είναι, μπορεί να γίνουν αποδεκτές. Έχω την ίδια άποψη με τον κύριο Σικλούνα και νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε μία διατύπωση η οποία θα μας επιτρέψει να δείξουμε την αποφασιστικότητά μας έτσι ώστε αυτός ο μηχανισμός να τεθεί σε εφαρμογή κάτω από καλές συνθήκες και να περάσει και το μήνυμα του Κοινοβουλίου. Δηλαδή ότι σε αυτή την περίοδο κλειδονισμών θα πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχουν μέτρα τα οποία μπορούν να προβληθούν έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ε, περιόδους κρίσης και τους οικονομικούς κύκλους που προβλέπονται. Ευχαριστώ πολύ. Ε, να ακούσουμε τους ε, εισηγητές ή όσους μιλούν εκ μέρους τους. Ε, εγώ έχω υποβάλει μια τροπολογία. Ευχαρίστω θα την αποσύρω. Ε, υπέρ της τροπολογίας 23. Ε, Απλά την υπέβαλα για να καταστήσω σαφές ότι έχω αντίρρηση σε κάποια μέρη του αρχικού κειμένου για τα οποία έχω μιλήσει ήδη. Ε, όμως θα αποσύρω την ε, τροπολογία μου για να μην εμπερδέψω το θέμα. Εκ μέρους της Άλντε, η Σίλβη. Ευχαριστώ. Εγώ κατανοώ αυτά που λέει ο Ζαν Πολ. Υπάρχει ένα θέμα δόγματος εδώ, δηλαδή τι κάνει το Κοινοβούλιο τη στιγμή που δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να αντιταχθούμε στη θέληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν θα είχε νόημα. Όμως το πρέπει να εκφράσουμε αυτό που θεωρούμε σωστό. Ακόμα και αν αυτή τη φορά δεν θα περάσει κάτι τέτοιο, δεν θα εισακουστεί. Γι' αυτό ήθελα να υποβάλω τροπολογίες έτσι ώστε να υπάρχει ένας αυτοματισμός στον όλο μηχανισμό. Θα μπορούσαμε να δεχτούμε ένα συμβιβασμό, αλλά για να επανέλθω σε αυτά που είπε ο Ζαμπόλ και εγώ ήρθα σε επαφή με τον ε, καθηγητή, με τον καθηγητή ο οποίος εκπροσωπούσε το, τα, τα κράτη σε επίπεδο συνταγματικού δικαστηρίου και νομίζω ότι πολλές φορές ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια κοινή ένωμη τάξη. Δηλαδή θα πρέπει να εκφράσουμε αυτό που θεωρούμε σωστό και να μην δεχτούμε μία μαξιμαλιστική προσέγγιση από ένα συνταγματικό δικαστήριο ενός κράτους μέλους. Ο Ραμόν θα προβάλλει αυτή τη θέση. Σας ευχαριστώ γιατί προσπαθήσατε να φτάσετε σε ένα συμβασμό, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να προβάλλουμε αυτή την ιδέα, ε, ακόμα και αν μας αγνοήσει το Συμβούλιο σε τελευταία ανάλυση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, όσον αφορά το άρθρο και την τροπολογία 23, εν μέρη καλύπτει αυτά που προτείνουμε και άλλωστε ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι οι συνθήκες να λένε τα πάντα. Μπορεί όμως να τις ερμηνεύσει κανείς με οποιοδήποτε τρόπο. Το πρόβλημα που έχω αυτή τη στιγμή είναι ότι βλέποντας τον τρόπο που αναπτύσσεται το θέμα αυτό της οικονομικής διακυβέρνησης, ε, τονίζεται ένα μέρος των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, μιλάμε κυρίως για την Γερμανία. Η Γερμανία θέλει η υπόλοιπη Ευρώπη να γίνει μια σειρά μικρών Γερμανιών. Δεν ε, θεωρώ ότι αυτός είναι ισορροπημένος ε, τρόπος προσέγγισης και γι' αυτό θέλουμε να τονίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μία σειρά στόχων που δεν εξυπηρετούνται από τον τρόπο που η Γερμανία και οι υποστηρικτές της ε, ερμηνεύουν τις συνθήκες και αυτό θέλουμε να διατυπώσουμε. Είναι πιο θολή η δική σας διατύπωση, καλύπτει όμως αυτό που προτείνουμε. Θα δούμε λοιπόν μήπως μπορούμε να στηρίξουμε τη συμβαστική σας τροπολογία. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Οι εξελίξεις ε, που βλέπουμε είναι ότι ε, παραπονιόμαστε εδώ και καιρό ότι η Γερμανία αποσύρεται από την Ευρώπη, τώρα βλέπουμε ότι επανέρχεται. Τώρα βλέπουμε όμως ότι αυτό γίνεται κυρίως για να ικανοποιήσει την επιθυμία της Γερμανίας για ε, νομική ασφάλεια. Ούτε ένας Γερμανός βουλευτής, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι παρόν στην συζήτηση αυτή. Αρχίζω λοιπόν να έχω κάποιες ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο που εξελίσσονται τα πράγματα. Είναι σοφό για τη Γερμανία να επιλέγει ανάμεσα σε δύο επιλογές, είτε να αποσύρεται είτε να υπαγορεύει. Νομίζω ότι ανάμεσα σε αυτές τις ε, δύο λύσεις ε, μπορεί να υπάρχει κάποια που να μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη συνένεση εντό Ευρώπη. Ε, φυσικά μπορούμε να μάθουμε καλά πράγματα από την Γερμανία, αλλά ο τρόπο που αντιμετωπίζει η Γερμανία το θέμα αυτή τη στιγμή Ε, μας οδηγεί στον κίνδυνο μιας αντίδρασης από τους ε, πολίτες ε, και τους, τους μη Γερμανούς πολίτες. Κάτι παρόμοιο που είδαμε το 2003 όταν οι Ηνωμένε Πολιτείες ξεκίνησαν πόλεμο κατά του Ιράκ και είχαμε ένα αίσθημα αντιαμερικανικό στην Ευρώπη και φοβάμαι ότι η αντιμετώπιση της Γερμανίας αυτή τη στιγμή θα οδηγήσει σε κάτι παρόμοιο. Δηλαδή αυτή η, η διάθεση θα οδηγήσει ε, ώστε ούτε τα καλά από τη, από γερμανική εμπειρία να μην γίνουν αποδεκτά από την υπόλοιπη Ευρώπη. Ε, αυτά ήθελα από του γερμανού Γερμανούς φίλους μου. Λυπάμαι πολύ που δεν είναι κανείς από αυτούς παρόν, αλλά έτσι είναι η ζωή. Ωραία, η Άστρη την επόμενη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ υπέβαλα μία τροπολογία σε αυτή την έκθεση Εγώ θέλω απλώς να προβάλλω μια διασάφηση, όχι να αμφισβητήσω το οτιδήποτε. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ο μηχανισμός σταθερότητας αφορά την Ευρωζώνη στο σύνολό της. Αυτό είναι σαφές. Αλλά και τα κράτη-μέλη ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια του ευρώ. Νομίζω ότι και ένας άλλος συνάδελφος υπέβαλε μία παρόμοια τροπολογία. Επίσης κάτι άλλο πιο σημαντικό θα πρέπει να διαγράψουμε αυτή την αλλαγή ερμηνείας από πλευράς Συμβουλίου του άρθρου 122 που επέτρεπε τη σύσταση του μηχανισμού σταθερότητας γιατί γνωρίζουμε ότι αυτή η, ερμηνεία είναι, αφορά καθαρά τον τραπεζικό τομέα αλλά δεν θα ήταν σκόπιμο να αποκλείσουμε την προσφυγή σε αυτό το άρθρο. Από νομικής πλευράς, το άρθρο 122 παραμένει ενισχύει. Δεν πρέπει να συγχαίουμε τα πάντα. Δεν μπορεί ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να είναι ο απότερος δικαστής των συνθήκων. Ξέρω ότι πολλές φορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίουμε τα πάντα. Ίσως ο Ζαν Πολ θα το κατανοήσει αυτό. Δεν θα πρέπει να τα κατατροπώνουμε όλα και να κινούμαστε με μία ρομφέα στο χέρι. Θα πρέπει να τηρήσουμε ένα μίνιμουμ κανόνων. Αυτό ήθελα να σας πω, να σας αιτιολογήσω δηλαδή, γιατί υπέβαλα την τροπολογία που γνωρίζετε. Um, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σάλλομ είναι ο τελευταίος ομιλητής στον κατάλογό μου. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος που θέλει να στήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι πρόσφατο μέλος αυτής της Επιτροπής, είμαι και αναπληρωτής στη θέση του Ερίκε Γκερέιρο και είμαι τακτικό μέλος της Επιτροπής Συνταγματικών Θεμάτων, η οποία τελικά θα αποφανθεί επί της ουσίας για τη μεταρρύθμιση των συνθήκων, διότι εδώ συζητούμε μια γνωμοδότηση της, ε, για μια γνωμοδότηση της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Θα ήθελα να τονίσω ότι έγιναν έντονες συζητήσεις στην Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων και γνωρίζουμε το ρόλο του Κοινοβουλίου σε αυτή τη μεταρρύθμιση της συνθήκης. Τη στιγμή που υπάρχει μία διακυβερνητική ολίσθηση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε μια κατάσταση βαθμίας αδυναμίας. Υπ' αυτή την έννοια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως είπε η κυρία Γκουλάρ, θα πρέπει να καταστήσει πρόδειλη τη θέση του, αναλαμβάνοντας μια διπλή ευθύνη. Καταρχήν, να προσέξουμε ως προς ενδεχόμενες μεταρρυθμίσεις που θα αφήσουν το αποτύπωμά τους σε μελλοντικές μεταρρυθμίσεις, δηλαδή δημιουργούμε ένα προηγούμενο. Τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη δραστηριότητα οικονομικής διακυβέρνησης που θα μπορούσε να σταθεί επικίνδυνη για το μέλλον και παράλληλα να μην μπορούμε να ανασχέσουμε αυτό που μας πρότεινε το Συμβούλιο να το ανασχέσουμε από πολιτικής πλευράς, γιατί πρόκειται για ένα επικίνδυνο μήνυμα έναντι των αγορών. Άρα, το πρώτο ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε. Το Συμβουλίο δεν είναι υποχρεωμένο να αλλάξει κάτι σε σχέση με μία γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου. Το Συμβούλιο μπορεί απλώς να συνεχίσει να προβάλλει τις δικές του θέσεις χωρίς να αλλάξει το περιεχόμενο της νομοδότησης. Όμως, δεν θα ήταν σκόπιμο να προτείνουμε αλλαγές και να μας αγνοήσει το Συμβούλιο. Τότε θα υπάρξει διάσταση απόψεων και θα, παραμέναν, θα παρέμεναν αδύναμες και οι δύο πλευρές από κάτι τέτοιο. Άρα θα πρέπει να βρούμε το δρόμο έτσι ώστε να καταστήσουμε πρόδειλη τη θέση μας, να πούμε ποιες είναι οι επιφυλάξεις μας στις προτάσεις του Συμβουλίου και επίσης να εξηγήσουμε τι θα θέλαμε να προωθηθεί πολύ περισσότερο σε επίπεδο οικονομικής διακυβέρνησης και τι συνταγματικές επιπλοκές θα είχε σε αυτή την περίπτωση. Το κρίσιμο όμως σημείο είναι το εξής. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο τοποθετούμε τις σκέψεις μας στην αιτιολογική σκέψη, στα εκτιμώντας δηλαδή προβάλλοντας τις επιφυλάξεις μας ή θα αλλάξουμε τις διατάξεις του κειμένου που μας απέστειλε το Συμβούλιο. Και μέσα στα πλαίσια των διατάξεων θα πρέπει να δούμε κατά πόσο δεχόμαστε μια νέα παράγραφο όπως μας απέστειλε το Συμβούλιο ή ένα νέο σημείο μέσα στο 136 που θα υποβληθεί βάσει τροπολογιών. Ποιο είναι το πρόβλημα με την εισαγωγή ενός νέου σημείου στο 136 και όχι της εισαγωγή μιας νέα παραγράφου. Το πρόβλημα έγκυται στο εξή. Ο μηχανισμός σε μία περίπτωση είναι διακυβερνητικό και στην άλλη πλευρά είναι κοινοτικό, ενδοκοινοτικός. Εάν λοιπόν μετατραπεί σε ενδοκοινοτικό, δηλαδή ξεχωριστή επιλογή, τότε υπάρχουν επιφυλάξεις ή ε, πολιτικές αμφιβολίες από πλευράς Γερμανίας και Ηνωμένου Βασιλείου, διότι το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρεί ότι δημιουργούνται νέες αρμοδιότητες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να διενεργηθεί δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως υπάρχει και μία άλλη σκέψη που είναι η ποσοτική διάσταση του μηχανισμού οικονομικής σταθερότητας, που θα μπορούσαν να εκφράσουν άλλοι καλύτερα από μένα. Δηλαδή, εάν υπάρχει μεγαλύτερη διάσταση από την παρούσα για να μπορέσει να δράσει προληπτικά και να μην ανταποκριθούμε σε μία μεγάλη κρίση, δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Θα πρέπει να μιλήσουμε για εισφορές κρατών μελών σε αυτή την περίπτωση. Άρα μετατρέπεται σε διακυβερνητικό το θέμα. Άρα τη στιγμή που αξιολογούμε τις διάφορες ε, τροπολογίες, θα πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσο θέλουμε έναν διακυ... όχι εάν θέλουμε ένα διακυβερνητικό μηχανισμό ή ενδοκινοτικό, αλλά αν θέλουμε ένα μηχανισμό σταθερότητας, χρηματοοικονομικής σταθερότητας ή όχι. Διότι ξέρετε ότι η μία προσέγγιση δεν θα γίνει αποδεκτή από το Συμβούλιο, ενώ η διακυβερνητική προσέγγιση θα αποδώσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα απαρνηθούμε ορισμένες πτυχές της ε, χρηματοοικονομικής σταθερότητας που θα μπορούσαν να έχουν συνταγματικό αντίκρισμα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και συνετοί στις τροπολογίες που θα υποβάλουμε και θα εγκρίνουμε. Και δέχομαι και τη συνετή και προσεκτική στάση των δύο εισηγητών. Θα προσπαθήσουν να φτάσουν σε μια συνενετική θέση που θα εκφράζει συνολικά τη θέση της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ. Ναι, ένα σχόλιο για τα όσα είπατε. Όλοι θα πρέπει να δεχθούμε ότι ορισμένοι τομεί θα παραμείνουν στην διακυβερνητική συνεργασία και δεν νομίζω ότι αυτή η αλλαγή τη συνθήκη θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως αφορμή ή ως παράθυρο που επιτρέπει να μπει περισσότερη διακυβερνητική συνεργασία, κάτι που ήδη βλέπουμε. Αυτό που υπερασπίζεται η παρούσα επιτροπή είναι η θέση του Κοινοβουλίου για θέματα όπως η πολυμερής εποπτεία. Σχετικά με το πότε, πώς και ούτω καθεξής θα αρχίζουν να λειτουργούν αυτοί οι μηχανισμοί. Ο, ο Ζητώ συγγνώμη, ήρθα με καθυστέρηση γιατί είμαι και σε άλλη επιτροπή όπου επίσης συζητούνται σημαντικά θέματα. Τώρα, για τα θέματα αυτά εδώ, εγώ είχα ζητήσει με τροπολογία στην δεύτερη φράση που λέει θα μείνουμε μόνο στην ουσία ή θα μπούμε και στις ε, κατατεθείς τροπολογίες. Εγώ του ελάχιστον θα έλεγα η δεύτερη φράση για τις ε, κρατικές ενισχύσεις δηλαδή που θα πρέπει να, είναι, να υπόκειται σε αυστερή αρεσιμότητα αυτό να διαγραφεί γιατί η συνθήκη της Λισαβόνας είναι κατά κάποιο τρόπο το σύνταγμα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Εγώ νομίζω ότι δεν εντάσσεται τέτοια ρύθμιση σε συνταγματικό κείμενο. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να μπει σε νόμο εφαρμογής, αλλά όχι στο ίδιο το συνταγματικό το εισαγωγικών κείμενο. Άρα θα πρέπει να φύγει αυτή η φράση. Αυτό είναι και το πρόβλημα που με απασχολεί περισσότερο. αν προσπαθήσω να βάλω το θέμα αυτό σε κάπως διαφορετικό πολιτικό πλαίσιο, πάντοτε γινόταν η συζήτηση για την Ευρώπη των δύο ταχυτήτων. Εάν βάλουμε αυτή τη φράση εδώ, στην ουσία αυτό κάνουμε. Προδιαγράφουμε μια Ευρώπη των δύο ταχυτήτων χωρίς να έχει καν συζητηθεί. Θα υπάρχει η ομάδα ευρώ, ζώνη ευρώ δηλαδή, η οποία θα υπαγορεύει το τι θα γίνεται. Θα είναι λοιπόν οι πιο ισχυρέ ε, οικονομικά χώρε και θα υπάρχουν και οι υπόλοιπε εκτό. Χωρί λοιπόν καμία συζήτηση θα έχουμε φτιάξει, κατά τη δική μου γνώμη, στο συνταγματικό μάλιστα επίπεδο μια Ευρώπη των δύο ταχυτήτων. Αυτό λοιπόν κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να γίνει. <clears throat> Τουλάχιστον όχι εδώ, όχι έτσι. Και στην Επιτροπή Σούρε αυτή τη στιγμή που συζητείται η πολιτική συνοχή πρέπει να συνδυαστεί και θα συνδυαστεί με αυτή την αιρεσιμότητα. Ούτε λοιπόν το αντίθετο μπορεί να εγγραφεί εδώ στην συνθήκη της Λισαβόνας γιατί θα έχει συνέπειες επιπτώσεις σε άλλους τομείς πολιτικής της Ένωσης. Όπως είπε η Σάρον τώρα για τον ανταγωνισμό, την προηγούμενη εβδομάδα πρότεινε η Άγγελα Μέρκελ αυτό το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας και στην συζήτηση που γίνεται στην Ομοσπονδιακή Γερμανία μαθαίνω ότι υπάρχει ένα non-paper της Μέρκελ που πάει να φέρει το θέμα αυτό σε ένα παράλληλο κοινοβουλευτικό επίπεδο, το οποίο θα κρίνεται, το, αυτό το παράλληλο κοινοβουλευτικό επίπεδο θα είναι τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών μελών, τα οποία θα συνέρχονται τακτικά μέσα στο χρόνο και εκεί θα αποφασίζουν. Και αυτό παράλληλα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάει δηλαδή τώρα να οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Και μακροπρόθεσμα, επαναλαμβάνω, θα ανατραπεί η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα καταστραφεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μακροπρόθεσμα, αυτό ξαναλέω. Έχω την εντύπωση, Γερμανός είμαι, δεν είμαι βεβαίως μέλος της ΣΕΝΤΕΟΥ, αλλά μου φαίνονται εκπληκτικά αυτά τα πράγματα που ξεπηδούν μέσα από τη χώρα μου ως, θα έλεγα, αντιευρωπαϊκές κινήσεις. Εγώ αριστερός είμαι συχνά πολύ επικριτικός απέναντι στα όσα συμβαίνουν στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είμαι Ευρωπαίος και αντιτάσσομαι σε αυτά που πάει να προωθήσει τώρα η Ομοσπονδιακή Γερμανία. Εγώ νομίζω λοιπόν πρέπει να ληφθούν αυτά υπόψη όταν θα σκεφτούμε και θα αποφασίσουμε και θα κρίνουμε περί τίνος πρόκειται. Νομίζω ότι πρέπει πράγματι να ασκήσουμε κάποια επιρροή και να ανακόψουμε αυτές τις ε, πορείες. Στην Επιτροπή Προϋπολογισμών στην αρχή της εβδομάδας είχαμε επίσης το θέμα αυτό. Η συνάδελφος Τρίπελ των Πράσινων και βασιζόμενοι στι ε, εμπειρίες που είχαμε με το σύστημα SWIFT τον προηγούμενο χρόνο, όπου το κοινοβούλιο είπαμε δεν είναι σε συναπόφαση, αλλά καλείται να γνωμοδοτήσει. Εάν το κοινοβούλιο δεν γνωμοδοτήσει, τότε το Συμβούλιο δεν μπορεί να προχωρήσει. Εγώ θεωρώ ότι αυτή είναι μια ιδέα που θα πρέπει να καθίσουμε λίγο να τη σκεφτούμε, ώστε να ασκήσουμε κάποια επιρροή, ώστε να μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε αυτή την ε, ε, εξέλιξη, γιατί όπως είπα πάει να γίνει μια στροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό βλέπω. Σας ευχαριστώ. Άρα δηλαδή τότε η ΑΦΚΟ θα πρέπει να κρατήσει τη γνωμοδότησή της, να μην υποβάλει γνωμοδότηση. Επιθυμεί κάποιος από τους άλλους συγητές να λάβει το λόγο, ο Ζαμπόλιο ο Έντουαρτ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Άκουσα τις διάφορες παρεμβάσεις. Συμφωνώ με την Σιλβή. Ε, εδώ το Κοινοβούλιο πρέπει βέβαια να τοποθετηθεί, να, να εκφράσει αυτό που θεωρεί δίκαιο, χωρίς υπερβολές που δεν θα εξυπηρετούσαν τίποτα, αλλά για τα ουσιώδη θέματα θα πρέπει να τοποθετηθούμε. Και το γεγονός ότι ενδεχομένως να έρθουμε σε σύγκρουση με το Συμβούλιο Υπουργών ε, είναι ένα ενδεχόμενο. Εν πάση περιπτώσει δεν θα είναι και πραγματική σύγκρουση γιατί δεν θα αποφασίσουμε εμεί τελικά. Αλλά έχουμε την, ε, το δικαίωμα να εκφράσουμε διαφορετική άποψη. Εν προκειμένου ας αποφύγουμε τη σχιζοφρένεια αυτή που ε, έγκυται στο να μιλούμε διαρκώς ε, για τις αγορές που λειτουργούν από στιγμή σε στιγμή και εμείς παλεύουμε χρόνια για να φτιάξουμε ένα κείμενο το οποίο ποτέ θα ικανοποιήσει όλο τον κόσμο. Αυτό που έχει σημασία σήμερα είναι η ταχύτητα. Είναι κατεπίγουσες οι εξελίξεις. Είναι τελείως διαφορετικός ο χρόνος του νομοθέτη και ο χρόνος των αγορών. Αυτό που αναμένουν οι πολίτες είναι απαντήσεις απαντήσεις από την Ευρώπη. Οι περισσότεροι από εμάς άλλωστε πιστεύουμε στην Ευρώπη. Οι μακρές συζητήσεις για το νομικό περιεχόμενο έχουν και ένα αποτέλεσμα, δηλαδή ορισμένες χώρες μπορούν και ρυθμίζουν τα πράγματα όπως θέλουν, περιθωριοποιώντας οριστικά πλέον το Κοινοβούλιο. Διότι η διακυβερνητικότητα δεν είναι τα ε, το, το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ίσως παίζουν και ένα ρόλο τα εθνικά κοινοβούλια, όχι όμως το Ευρωπαϊκό. Άρα πρέπει να κάνουμε να ακουστεί η φωνή μας, να πάρουμε θέσεις ρεαλιστικές για τα κέρια θέματα της λειτουργίας της Ευρώπης. Και συμφωνώ με τον Γιούργεν που λέει ότι αυτό που τίθεται σε αμφισβήτηση εδώ είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Ευρώπη στο οικονομικό επίπεδο ίσως η διακυβερνητική συνεργασία να είναι αποτελεσματική και πιο αποτελεσματική από την κοινοτική συνεργασία και όπως μας έλεγε ο κ. Ρομπλές, παλαιός πρόεδρος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συχνά ξεκίνησε μια συνεργασία διακυβερνητικά για να καταλήξει να γίνει κοινοτική. Αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε να περάσει μια δεκαετία για τέτοια θέματα. Τα οικονομικά θέματα θίγουν την καθημερινή ζωή των πολιτών μας. Και γι' αυτό και με τον Έντουαρτ αναζητούμε διατυπώσεις και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε που θα επιτρέπουν και ρεαλιστές να είμαστε, να μην ζητάμε πράγματα παράλογα, αλλά και ταυτόχρονα να δείχνουμε καθαρά ποιε είναι οι επιθυμίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τι πιστεύουμε για τον μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων, την αλληλεγγύη στην ζώνη ευρώ, έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να εκφράσει με ρεαλισμό, ε, σοφία και σαφήνεια τις θέσεις του. Διότι εν τέλει οι μόνες μάχες που χάνει κανείς είναι οι μάχες που δεν διεξήγαγε ποτέ. Είδαμε τώρα και τα θέματα εποπτείας, όπου πριν από την συζήτηση θεωρούσαμε ότι το Συμβούλιο θα υιοθετούσε την δήλωση της Ουγγρικής Προεδρίας, υποστηρίζοντας έτσι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να έχουν αυτονομία οι εποπτικές αρχές. Εάν μπορούμε να, κάνουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε να προχωρήσουν τα πράγματα με ρεαλισμό και με τον Έντουαρτ σε συνεργασία αυτό κάνουμε, διατυπώνουμε τις σκέψεις που θα εκφράσουν με καλύτερο τρόπο. Τώρα γιατί ένα street ruling που προσέχω πάρα πολύ πάντοτε τα σοφά λόγια που λέει, όταν μου λέει ότι πρέπει να διαγράψουμε την παράγραφο αυτή. Εδώ δεν συμφωνώ απόλυτα, διότι οι χώρες μέλη αναγνωρίζουν ότι έχουν χρησιμοποιήσει τις παραγράφου αυτές, το άρθρο αυτό, για στόχους ξένους. Και λένε ότι από τη στιγμή που θα μπει σε ισχύ το 136.3 η γάμα, το 122 θα συνεχίσει να υπάρχει, αλλά θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για τους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκε, για την αλληλεγγύη δηλαδή απέναντι σε θεομηνίες και άλλες φυσικές καταστροφές. Δεν θα ξαναστρεβλώσουμε λοιπόν την ερμηνεία του άρθρου αυτού για να το κάνουμε λέει πράγματα που δεν λέει. Εγώ νομίζω λέω ότι τέλος πάντων δεν θα πω στα θρησκευτικά τώρα γιατί τα άλλοι τα ξέρουν καλύτερα, αλλά τέλος πάντων δεν θα είναι και κέριο ε, θέμα να το καταργήσουμε το άρθρο αυτό. Αλλά το λέω προς την Άστριντ για να έχει υπόψη ότι ό,τι και να λέει το σημειώνουν προσεκτικά οι εισηγητές. Τότε να κλείσουμε τη συζήτηση για τις τροπολογίες αυτές. Η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα στο Στρασβούργο. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή στην ε, ε, αρμόδια της Επιτροπή ε, μάλλον θα προγραμματιστεί άλλη μέρα, ήταν προγραμματισμένη για τις 14 Μαρτίου. Ε, κανονικά ήταν να πάει στην πρώτη ολομέλεια του Μαρτίου. Μπορεί αυτό να αλλάξει, μπορεί και όχι. Αλλά και καλό είναι να έχουμε υποβάλει εμείς τη γνωμοδότησή μας. Προχωράμε στο σημείο 5. Η δημιουργία μεταβατικών ρυθμίσεων ε, στα πλαίσια διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών. Ζων Πολ, νομίζω θα μιλήσει εσύ εκ μέρους του Ντέιβιτ Κάζα. Σωστά. Ναι, τον αντικαθιστώ. Αλλά μου δόθηκαν ορισμένες πληροφορίες πριν από την αρχή της συνεδρίασης και πρέπει να πω ότι είμαι λίγο χαμένος εδώ. Γιατί δεν τις βρίσκω αυτές τις σημειώσεις. Ακούτε, Désolé, Voilà. J'y suis. <coughs> Et eh non, c'est Edouard qui Ο Έντουαρντ είχε ασχοληθεί με το θέμα. Λοιπόν, ο κύριος Κάσας, ζητεί συγγνώμη που δεν είναι παρόν, αλλά έπρεπε να επιστρέψει στη Μάλτα για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του. Θα σας διαβάσω λοιπόν αυτά που έγραψε για να δείτε ποιες είναι οι θέσεις του εισηγητή ως προς διάφορες τροπολογίες. Ως προς τις διμερές επενδυτικές συμφωνίες υπάρχουν τροπολογίες, οι περισσότερες ε, έχουν στόχο να αποσαφωνήσουν το κείμενο. Δέχεται 32, 33, 35, 38 και 39 και θα συνεργαστεί με τους συγγραφείς συντάκτες έτσι ώστε να ενταχθούν στο κείμενο. Δέχεται το, την τροπολογία 31, την ειδική αυτή ε, ρήτρα, αλλά θέλει να δούμε καλύτερα την διατύπωση έτσι ώστε να έχουμε ένα ε, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα σε σχέση με τις ε, επενδυτικές συμφωνίες, διεθνείς επενδυτικές συμφωνίες, πολλές τροπολογίες είναι επικοδομητικές. Δέχεται αυτές τις τροπολογίες και εργάζεται για να ενταχθούν πολλές από αυτές τις ε, τροπολογίες συμβασμού. Είναι υπέρ των διότι δεν υπάρχει αναγνωρισμένος ορισμός των άμεσων αλλοδαπών επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ των 2, 4, 8, 10 και 15 για να αποσαφινιστεί το κείμενο. Γνωρίζει ότι ορισμένοι συνάδελφοι θεωρούν ότι μία πολιτική επενδύσεων θα πρέπει να ενθαρρύνει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στα πλαίσια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, των, και της προστασίας του περιβάλλοντος. Θεωρεί ότι είναι ένας πολύ εύλογος στόχος και θα προσπαθήσει να βρει τις σωστές διατυπώσεις στο κείμενο. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι οι άμεσες ε, επενδύσεις της αλλοδαπής θα πρέπει να την χάνουν υποστήριξη ακόμα και σε χώρες που δεν συμμερίζονται αυτές τις αξίες. Ο κύριος Κάζα θα ήθελα να ευχαριστήσει όλους τους συναδέλφους που συνεισέφεραν στην σύνταξη του κειμένου και ελπίζει το τελικό έγγραφο να είναι συνενετικό στα πλαίσια της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σκιώδης. Ίσως μπορώ να εκφραστώ στα γαλλικά, όπως και ο προλαλής σας. Ως προς τις τροπολογίες θα ήθελα να αποβαλω δυο δύο-τρία σχόλια ως προς τις δικές μου τροπολογίες. Πιστεύω ότι είναι καθήκον μας να λάβουμε υπόψη τη συνθήκη, δηλαδή να έχουμε συνενετικές πολιτικές για να φτάσουμε στους στόχους της συνθήκης. Άρα οποιαδήποτε αλλοδαπή δράση εμπορίου, γεωργίας και ούτω καθεξής θα πρέπει να συνάδει με τους στόχους μας, δηλαδή τη μείωση της φτώχειας ανά τον κόσμο. Αυτό βεβαίως ε, ενυπάρχει στις συνθήκες και πρέπει να το σεβαστούμε αλλά για τις ε, διμερείς επενδύσεις θα ήταν σκόπιμο να προσδιοριστεί. Ως προς τον ορισμό των άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό υπάρχει μία τροπολογία που διευκρινίζει καλύτερα αυτό το πλαίσιο, αλλά νομίζω ότι δεν είναι σκόπιμο κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι η πρόταση της Κομισιόν αρκεί, η πρόταση ορισμού ιδιαίτερα ως προς τα χαρτοφυλάκια, της υπό υπομορφή χαρτοφυλακίων που αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα δεν μπορούμε να τις αποκλείσουμε από το κείμενο. Όταν μιλάμε για dispute settlements, για διακανονισμούς μέσα στα πλαίσια διαφορών, στα πλαίσια του ΠΟΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλόμενο μέρος, διότι πρόκειται για αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα νομίζω ότι δεν πρέπει με τις τροπολογίες να πούμε ότι μόνο εκεί όπου κρίνουμε σκόπιμο η Επιτροπή συμμετέχει στη διαδικασία. Δηλαδή εκεί όπου υπάρχει διαφορά νομίζω ότι η Επιτροπή πάντα πρέπει να συμμετέχει στη διαδικασία. Δεν συμφωνώ με αυτή την τροπολογία. Αυτά. Και σας ευχαριστώ. Fine. Um... Ωραία. Υπάρχει κανείς που θέλει να πάρει το λόγο? Τότε να προχωρήσουμε στην επόμενη έκθεση του κυρίου Κάζα. Σημείωσα τις παρατηρήσεις σας και θα ήθελα, θα τις διαβάσω τον κύριο Κάζα και να τον συγχαρείτε για το κείμενο. Να ακούσουμε τους σκιώδεις εισηγητές για την δεύτερη ε, έκθεση Κάζα, η μελλοντική ευρωπαϊκή πολιτική διεθνών επενδύσεων. Είναι παρόν ο Ραμόν, όχι. And Ούτε ο Νομίζω μπορούμε τότε να κλείσουμε και τις δύο εκθέσεις. Κύριε Κοζέ, νομίζω ότι τελείωσαν οι σημειώσεις σας. Όπως και να έχει, ας κοιτάξουμε το χρονοδιάγραμμα. Διαβάζω το τις σημειώσεις εξέταση των τροπολογιών. 10 Φεβρουαρίου. Ψηφοφορία στην Επιτροπή ΕΚΟΝ 28 Φεβρουαρίου. Ε, ψηφοφορία στην ΕΝΒΗ που είναι αρκόδια ψηφουσία στις 3 Μαρτίου. Ολομέλεια ε, τον Απρίλιο. Θα πάει στην πρώτη Ολομέλεια του Απριλίου. Fine. We will be, uh, Θα κάνουμε ένα διάλειμμα λίγων λεπτών. Παρακαλώ παραμείνετε στην αίθουσα. Θέλουμε... Και παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε την ε, κάρτα σας για τις ψηφοφορίες, γιατί έχουμε μία ψηφοφορία. Μπορούμε να συνεχίσουμε.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 διάλειμμα μισή ώρας, πρέπει όμως να έρθετε για την ψηφοφορία. Και θα πρέπει να έχουμε απαρτία για την ψηφοφορία. Σας παρακαλώ λοιπόν να έρθετε στις 11.30. Señorías, señorías, vamos a dar continuación a la Έχουμε μια ψηφοφορία αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, μια γνωμοδότηση δηλαδή της Επιτροπής μας που θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εξουσίας Επιτροπή Απασχόλησης για θέματα απασχόλησης των χωρών μελών. Έχετε μπροστά σας την λίστα ψηφοφοριών. Τροπολογία 1 του εισηγητού. Παρακαλώ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα. Παρακαλώ πάρτε τις κάρτες σας, όσοι τις έχετε και όσοι δεν έχετε να το ανακοινώσετε στη γραμματεία για να το λάβουμε υπόψη μας. να Προτείνουμε την πρόταση ψηφίσματος. Υπέρ παρακαλώ, διακόπτη ο Προεδρεύων. Με ανάταση του χεριού, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να συγχαρώ τον εισηγητή πέρα της ψυχοφορίας. Τώρα περνάμε στην έκθεση του κυρίου Κλίντς για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Κύριε Κλίντς, έχετε το λόγο. Καλά, δεν πειράζει, θα τα πω στα γερμανικά. Γιατί είναι παρόντες οι διερμηνείς και θέλω να τους επιτρέψω να εργαστούν σκληρά. Ευχαριστούν οι διερμηνείς τον Πρόεδρο. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω όλους και όλους τους συναδέλφους που έχουν καταθέσει τροπολογίες για την έκθεσή μου ιδίας πρωτοβουλίας για τους οργανισμούς κρίσης πιστοληπτικής ικανότητας, περίπου 200 τροπολογίες. Μεγάλος αριθμός των τροπολογιών αυτών οφείλεται στο ότι έγιναν κατ' επανάληψη διάφορες ε, τροποποιήσεις και είδα επίσης ότι υπάρχει και μια σχετικά ευρία συνένεση για, πολλά, για πολλές από τις παραγράφους, όχι για όλες βέβαια. Σε ένα από τα θέματα έχουμε ωστόσο απόκληση απόψεων, το θέμα δηλαδή εάν και κατά πόσον θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός οργανισμός για να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των ε, ε, οργανισμών αυτών, των οίκων αυτών. Θα έρθω όμως σε λεπτομέρειες. Μαζί με τους και ηγητές έχουμε διεξαγάγει τον Φεβρουάριο μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και βάλαμε τις βάσεις για την εργασία μας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα μπορέσουμε να υποβάλουμε κάποιες συμβιβαστικές ε, προτάσεις στους συναδέλφους. Τώρα, πού βρισκόμαστε λίγο μετά πλέον από την εξέταση των ε, τροπολογιών. Σε ό,τι αφορά τώρα τον οργανισμό αυτό, εκεί πραγματικά οι απόψεις διήστανται. Αφενός έχουμε μια πρόταση της ομάδας ECR, η οποία αμφισβητεί ολόκληρο το μοντέλο αυτό. Εγώ συναντήθηκα με τον κύριο Άσχολη Φόξ πριν από δύο ημέρες και μετά από την συζήτηση που διεξήγαγα μαζί του, μου δημιουργείται η εντύπωση ότι δεν αποκλείει πλέον απολύτως ε, το Ίδρυμα αυτό. Θέλει κάτι το οποίο βεβαίως πάντοτε εγώ υπεστήριξα, δηλαδή εάν καταναλωθεί το κεφάλαιο του οργανισμού αυτού να, και να μην μπορεί να σταθεί μόνο του στα πόδια του, να ε, επαναχρηματοδοτηθεί. Όχι, και εγώ αυτό θέλω. Να είναι ουδέτερη χρηματοδότηση. Στον οργανισμό αυτό θα είναι, όπου θα είναι απολύτως ανεξάρτητος και ουδέτερος, δεν θα μπαίνει μέσα ούτε πολιτικός ούτε ε, τίποτε άλλο στην διοίκησή του. Και εφόσον το κεφάλαιο του Ιδρύματος νομίζω θα χρειαστεί με μια περίοδο τριών έως τεσσάρων ετών μέχρι να μπορεί να σταθεί μόνο του το Ίδρυμα αυτό, ο οργανισμός αυτός, να μην θεωρήσει ότι εφόσον έχει αναλωθεί το κεφάλαιο αυτό θα επαναχρηματοδοτηθεί. Είτε θα τα καταφέρει να σταθεί μόνο στο οργανισμό είτε όχι. Υπό τι προποθέσει αυτέ νομίζω ότι ο κ. Άσουλη Φόξ δεν είναι πλέον τόσο αντίθετο. Εξ τώρα από άλλε πλευρέ και κυρίω από του σοσιαλδημοκράτε και βεβαίω και από την ενωτική αριστερά αλλά και από τους πράσινους νομίζω υπάρχουν απόψεις που λένε ότι θα πρέπει να είναι δημόσιος ο οργανισμός αυτός, rating agency, και θα πρέπει να υπαχθεί de facto στο ελεγκτικό συνέδριο. Εκεί όμως εγώ αντιμετωπίζω, πώς να πω, έχω σοβαρές αντιρρήσεις. Πρώτον, δημόσιος οργανισμός κρίσεως ε, πιστοληπτικής ικανότητας δεν θα είναι τόσο ανεξάρτητος όσο θα πραγματικά θα θέλαμε και όσο πρέπει να θέλουμε να είναι απόλυτα ανεξάρτητος δεν θα είναι ένα τέτοιο οργανισμό και αξιόπιστο στι αγορέ, αν δεν είναι απόλυτα ανεξάρτητο. Εφόσον είναι δημόσιο οργανισμό αυτό, ασφαλώ θα καλυφθεί η σύνθεση των συμβουλίων του κτλ. με άλλα κριτήρια, με κριτήρια πολιτικά. Δεν ξέρω. Θα είναι πολύ προβληματικό αυτό. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, τίθεται το ερώτημα πώς θα στελεχωθούν οι εποπτικές αρχές η κυβέρνηση, ο κ. Σαρκοζή είπε ότι θέλει να του ορίσει, να ορίζει η κυβέρνηση. Αυτό προκαλεί σημαντικότατε επιφυλάξει για να μην πω ότι και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αντίθετη, διότι οι εποπτικέ αρχές οφείλουν να είναι απολύτω ουδέτερε. Κάτι τέτοιο λοιπόν θα ήταν βλαβερό για τον οργανισμό αυτό κατά τη γνώμη μου. Όσον αφορά όσον αφορά το ελεγκτικό συνέδριο, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Δεν υπάρχει νομική βάση να θεωρηθεί αρμόδιο το ελεγκτικό συνέδριο. Τα καθήκοντα του ελεγκτικού συνεδρίου είναι απολύτω σαφώ καθορισμένα. Σύμφωνα με τις συνθήκες δηλαδή, ελέγχει όλα τα έσοδα και τις δαπάνες των ε, ευρωπαϊκών κοινοτήτων, της Ένωσης και ούτω καθεξής. Κατά τα λοιπά, δεν υπάρχει περιθώριο για ανάληψη άλλων δραστηριοτήτων. Θα επανέλθω για το ενδεχόμενο να έχει ένα ιδιαίτερο ε, ρόλο το ελεγκτικό συνέδριο στα λεγόμενα sovereign debts. Αυτά τώρα για τον οργανισμό αυτό. Τώρα, για το να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός, να συντονιστούν ε, περιφερειακώς δρόντες οργανισμοί πιστοληπτικής ικανότητας σε ένα ενιαίο, κάτω από μια ενιαία ευρωπαϊκή ομπρέλα. Αυτό όμως θεωρούν πολλοί και εγώ ότι δεν θα είναι επαρκώς διαφανές και αντικειμενικό. Θα χρειαστεί να ξανασυζητηθεί λοιπόν με του ε, συναδέλφους αυτό. Εγώ θεωρώ εν πάση περιπτώσει ότι ορισμένε προποθέσει μπορεί να ε, λειτουργήσει, αν και δεν θα πρέπει να έχουμε ψευδεστήσει. Οι φυστάμενοι οργανισμοί, οι οποίοι δρούν μονάχα εθνικά ή περιφερειακά, είναι πάρα πολύ εξειδικευμένοι. Έχουν εξειδικευθεί σε περιορισμένου τομεί ή σε περιορισμένο τομέα. Εξετάζουν, α πούμε, μόνο πιστοποιητικά ή κάνουν rating μονάχα για μια χώρα ή για ορισμένε χώρε και να τους φέρουμε τώρα να δράσουν αποτελεσματικά σε ένα διεθνές επίπεδο δεν θα είναι πολύ απλό ούτε θεωρώ ότι για παράδειγμα από 10 χώρες συνέρχονται τώρα 10 οργανισμοί και ενώνουν τις ε, δραστηριότητές τους ότι θα μπορούν ξαφνικά να καλύψουν ολόκληρο το φάσμα που καλύπτουν μεγάλη παγκόσμια οίκη και να είναι ανταγωνιστές μαζί τους. θα πρέπει να γίνονται, λέμε μετά, δύο υποχρεωτικά rating για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, για τα διαφρομένα προϊόντα. Είπαμε λοιπόν ότι αφενός ο εκδότης, ο issuer, θα πληρώνει δύο rating, τον ένα οργανισμό θα τον επιλέγει μόνος του, τον δεύτερο δεν θα τον επιλέγει ο ίδιος, για να υπάρχει η διασφάλιση ότι δεν θα υπάρχει μεγάλη ε, σύμπτωση συμφερόντων μεταξύ Ίσουερ και... Αλλά μπορεί να το κάνει η ΕΣΜΑ για παράδειγμα. Εδώ οι πράσινοι προτείνουν να μην γίνει αυτό μονάχα για ορισμένα διαρθρωμένα προϊόντα, αλλά καταρχήν να καλύπτονται όλα τα προϊόντα που πρόκειται να ε, αξιολογηθούν. Εγώ βρίσκω ότι αυτό είναι κάπως υπερβολικό. Πρέπει να εξετάσουμε τη σκοπιμότητά του, διότι κάπου αλλού λέμε ότι έχουμε την εντύπωση ότι οι rating agencies επιβάλλεται δηλαδή η δραστηριότητά τους σε υπερβολικά πολλές ε, περιπτώσεις. Και αυτό ισχύει και για τα δημόσια χρέη, τα οποία προ δεκαετιών, προ 25-30 ετών, σε πολλές περιπτώσεις, το δημόσιο χρέος δεν υφίστατο rating από rating agencies. Πήγαινε λοιπόν στις ε, αγορές, το δημόσιο χρέος, και αγοράζονταν ή όχι από τους επενδυτές χωρίς rating. Τώρα δεν υπάρχει πλέον αυτό και πολλοί θεσμικοί επενδυτές, εταιρείε κλπ. υποχρώνονται και από το καταστατικό τους και από την ισχύουσα νομοθεσία να επενδύουν μοναχά σε προϊόντα τα οποία διαθέτουν ένα ελάχιστο rating. Εδώ λοιπόν πρέπει να τεθεί το ερώτημα μήπως θα πρέπει να επιβάλλουμε την υποχρέωση στους ίδιους τους θεσμικούς επενδυτές να κάνουν ένα μέρος του rating και αν σκεφτώ για παράδειγμα την περίπτωση μεγάλων συνταξιωτικών ταμείων ή άλλων τέτοιων πολύ μεγάλων οργανισμών, μπορούν να κάνουν τη δουλειά αυτή μόνοι τους. Και για την αξιολόγηση δημόσιου χρέους, όλες οι πληροφορίες που χρειάζεται κανείς για να κάνει το rating είναι διαθέσιμες, είναι δημόσιες είτε μέσω των στατιστικών, είτε μέσω των κεντρικών τραπεζών και ούτω καθεξής. Είναι λοιπόν όλα αυτά διαθέσιμα και μάλιστα και ε, πάρα πολύ επικαιροποιημένα. Άρα δεν υπάρχει πραγματικά λόγος να γίνεται πάντοτε αναφορά στα προϊόντα των τριών μεγάλων ε, οίκων. Υπάρχει και η πρόταση των σοσιαλδημοκρατών το, το ελεκτικό συνέδριο να αναλάβει την κρίση του sovereign debt. Εγώ το θεωρώ αυτό λίεν ρηψοκίνδυνο, διότι δεν εξασφαλίζεται πλέον ε, αντικειμενική αξιολόγηση, διότι είναι μοιραίο να υπάρξουν πολιτικές επιρροές και γι' αυτό νομίζω δεν μπορεί να γίνει. Ένα θέμα ακόμη που είναι ιδιαίτερα αμφισβητούμενο το θέμα της ευθύνης. Το εξετάζω αυτό διότι οι μεγάλες rating agencies παριστάνουν δήθεν ότι το μόνο που κάνουν είναι να εκφράζουν μια γνωμοδότηση. Λένε ότι εμείς δεν λέμε παρά μόνο τη γνώμη μας. Και ο καθένας μπορεί ελεύθερα να εκφράζει τη γνώμη του και γι' αυτό στην πραγματικότητα δεν έχει καμία συνέπεια. Αλλά De facto τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Κάθε κράτος έχει, διαθέτει ένα αστικό δίκαιο και σύμφωνα με το αστικό δίκαιο μπορεί κανείς να προσφύγει στα δικαστήρια εφόσον υπάρχει αμέλεια και να ζητήσει επιβολή κυρώσεων. Αυτό ισχύει και για τα rating agencies. Όμως οι ρυθμίσει είναι τόσο διαφορετικές ανάμεσα από χώρα σε χώρα μάλλον ώστε δεν μπορεί να ισχυριστεί κανεί ότι στην Ευρώπη έχουμε μια κοινή προσέγγιση. Η πρόταση λοιπόν είναι η Κομισιόν τουλάχιστον να εξετάσει εάν μπορούμε να προχωρήσουμε προς κάποια κατεύθυνση ώστε τουλάχιστον σε περίπτωση βαριάς αμέλειας, gross negligence, να μπορεί να διαπιστωθεί ευθύνη. Δεν πρόκειται βέβαια για να ε, καταστήσουμε υπόλογη μια rating agency επειδή εκ των υστέρων η άποψή της αποδείχθηκε ότι ήταν ορθή ή όχι, δεν έχουν και καμιά κρυστάλλινη σφαίρα και αυτοί για να ξέρουν τι θα γίνει στο μέλλον. Μπορεί κάποια στιγμή μία από τις αξιολογήσεις τους αυτές να αποδειχθεί ότι δεν ήταν σωστή. Αλλά αυτό που απαιτείται είναι τα κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιούν να είναι απόλυτα αξιόπιστα και επιστημονικά ποιοτικά. Και εδώ εγώ έχω σοβαρές επιφυλάξεις όταν σκέφτομαι για παράδειγμα τα ratings των διαθρωμένων προϊόντων που είχαν ε, σχέση με τις επιστώσεις subprime όπου κατά εκατοντάδες τα, αν μη χιλιάδες τα διαθρωμένα προϊόντα πέρασαν από το rating ταχύτατα και ακόμα και οι ίδιοι εκπρόσωποι των ε, οργανισμών πιστοληπτικής αξιολόγησης δέχονται ότι ίσως τότε να μην είχαν γίνει τα πράγματα τόσο ε, επαγγελματικά ή σε τέτοιο επίπεδο αξιοπιστίας όπως θα έπρεπε. Και σε τέτοια περίπτωση θα έπρεπε να είναι υπόλογοι. Τώρα ποιο θα είναι υπόλογο, ποιο θα μπορεί μάλλον, θα μπορεί μάλλον να προσφύγει εναντίον του, δεν μπορούμε να ε, θεωρήσουμε ότι ο κάθε επενδυτή, ο τελευταίο επενδυτή θα μπορέσει να του σύρει στα δικαστήρια. Θα μπορούσαμε να, να το δούμε το ενδεχόμενο αν ίσως η ΕΣΜΑ θα μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα. Να εξετάσει δηλαδή αν υπάρχει περίπτωση βαριάς αμέλειας και ενδεχομένως να ε, κληθεί να αναλάβει δράση. Λιγότερο αμφιλεγόμενα είναι ε, θέματα του level playing field πρόσβαση στι πληροφορίες. Υπάρχουν και εδώ πάρα πολλές τροπολογίες που νομίζω ότι μπορούμε να τις συγχωνεύσουμε σχετικά εύκολα σε συμβιβαστικά κείμενα. Αυτές που είναι πιο κριτικές τις έχω ήδη εξηγήσει. Η συνεργασία μου και με τους πιο ηγητέ και με την Κομισιόν ήταν καλή. Η Κομισιόν ήθελε να καταλήξει στην πρότασή της ήδη πριν από το καλοκαίρι, τώρα φαίνεται μάλλον να οδεύει προς Σεπτέμβρη. Θα κάνουμε και άλλη συνάντηση με τους πιο ηγητέ στις 2 Μαρτίου για να συζητήσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμά μας ώστε να ψηφίσουμε στις 16 Τρίτου στην Επιτροπή ΕΚΟΝ και αυτό μάλιστα είναι και επίγον σιγά σιγά διότι η, ε, η μου η οποία ασχολείται ιδιαίτερα με το θέμα αυτό θα γεννήσει το γιο της τρεις εβδομάδες μετά από την ημερομηνία αυτή. Ε, Ευχαριστούμε Κύριε Κλίνς, θα δώσουμε το λόγο στους ε, σκιώδες. Καταρχήν στον Ζαν Πολ Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητέ Βόλφ, νομίζω ότι θα πρέπει να... Μάλλον, ε, ελπίζω να τα καταφέρει ο βοηθός σου μέχρι τέλους, όπως η δική μου, η οποία τα κατάφερε πολύ καλά, δούλεψε μέχρι τέλους και έχει ένα μικρό γιο που φέρει το όνομα Αντουάν. Μπάς περιπτώσει, θα επανέλθω σε δύο-τρία ζητήματα που έθιξες. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι η δραστηριότητα πιστοληπτικής ικανότητας είναι μια καθαρά εμπορικού χαρακτήρα ιδέα. Και θα ήθελα να πω ότι δεν θα είχε νόημα να αποκλείουμε και δημόσιους οργανισμούς. Δηλαδή, είτε θα μιλάμε για δημοσίους υπαλλήλους είτε όχι. Το θέμα αυτό είχε φυγεί το 2009 κατά το πρώτο τμήμα σύνταξης ε, αυτού του κανονισμού και πολλές ιδέες απομακρύνθηκαν. Τώρα, Ως προς τον οργανισμό αυτό έχω αμφιβολίες, γιατί δεν καταλαβαίνω πώς θα μπορέσει να ενταχθεί εδώ. είτε υπάρχει ε, μία νομική εμβέλεια την οποία δεν γνωρίζουμε, δηλαδή θα πρόκειται για ένα νομικό πρόσωπο αλλά με βάση αυτά που είπες, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς θα έχουμε μια, έναν τέταρτο οργανισμό πιστοληπτικής ικανότητας που θα διαδραματίσει τον ίδιο ρόλο με τους άλλους. Δηλαδή θα έχουμε εισαγάγει ορισμένα στοιχεία για να εξασφαλίσουμε την ανεξαρτησία, τον επαγγελματισμό και ούτω καθεξής. Δεν με ενθουσιάζει η ιδέα εξορισμού, αλλά η τροπολογία μου αφορά τη διενέργεια μιας μελέτης αντικτύπου. Θυμόσαστε ότι στην προηγούμενη θητεία ένα συνάδελφος ασχολήθηκε με τη σύσταση μιας, ε, ενός οργανισμού πιστοληπτικής ε, ικανότητας και μας είχε ορίσει τις κεφαλαιοχικές ανάγκες ενός τέτοιου οργανισμού για την ίδρυσή του. Ως προς τη διπλή βαθμολογία θα μπορούσα να πω ότι συμφωνούμε και εμείς. Θα ήθελα όμως να λάβω υπόψη ε, μία διατύπωση η οποία λέει ότι θα πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτούς τους οργανισμούς, να αποτοξινωθούμε από οργανισμούς πιστοληπτικής ικανότητας. Αυτό είχε πει ο πρόεδρος των ε, γαλλικών κινητών αξιών. Θα πρέπει λοιπόν να μας απασχολήσει αυτό το θέμα. Κάποια μέρα ίσως θα πρέπει να διαγράψουμε αυτό τον ε, υποχρεωτικό χαρακτήρα. Και να υπάρχουν εμπορικοί οργανισμοί που να βαθμολογούν γιατί η παρούσα κατάσταση δεν είναι καθόλου ικανοποιητική. Οι οργανισμοί αυτοί διαδραματίσουν ένα ρόλο, αλλά το ίδιο κάνουν και οι επενδυτές όταν αναλαμβάνουν ορισμένους κινδύνους. Το γεγονός ότι ο βαθμός επηρεάζει τις κινητές αξίες, αυτό ε, αφορά το γεγονός ότι πολλοί επενδυτές εξαρτώνται άμεσα από τους οργανισμούς αυτούς. Γι' αυτό και ο Ζουγιέ είχε αναφέρει ότι θα πρέπει να αποτοξινοθούμε από τους οργανισμούς πιστοληπτικής ικανότητας. Εν πάση περιπτώσει θα, έχουμε, θα προβάλλουμε στοιχεία συμβιβασμού που ελπίζουμε να λάβει υπόψη η Κομισιόν. Η Άννη Ποδηματά το λόγο. Uh, President. Thank you. Uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ, κύριε Κλίνς, για την ε, παρουσίασή σας. Εξ του κυρίου Πιτέλα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη μέχρι τούδε εργασία σας. Θα ήθελα να υποβάλω ορισμένα σημεία που σχετίζονται με το προσχέδιο έκθεσή σας. Το πρώτο σχετίζεται με το γεγονός ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ρυθμιστικό σύστημα βασίζεται σε αυτές τις βαθμολογίες για ρυθμιστικούς σκοπούς. Ο κύριος Πιτέλα πιστεύει ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιόν καταρχήν να αναθεωρήσει και να δει πώς τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν τις βαθμολογίες για ρυθμιστικούς σκοπούς και δεύτερον να λάβουμε υπόψη την ε, δική σας πρόταση για να έχουμε δύο βαθμολογίες σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο κύριος Πιτέλα προτείνει ότι μία από τις δύο βαθμολογήσεις θα πρέπει να προέρχεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ε, Βαθμολόγησης και είπατε στην εισήγησή σας ότι θα πρέπει να ζητήσουμε τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού οργανισμού βαθμολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που θα ασχολείται με όλους τους τομείς ε, βαθμολόγησης. Πιστεύουμε λοιπόν ότι υπάρχει συνένεση ως προς το γεγονός ότι υπάρχουν ε, ξεχωριστά προγράμματα και δεν υπάρχει λογοδοσία από την άλλη. για τον τρόπο του πώς λειτουργούν τρεις οργανισμοί πιστοληπτικής ικανότητας. Σε σχέση με το δημόσιο χρέος, κάνατε ορισμένα σχόλια και νομίζω ότι αυτό που φαίνεται στην τρέχουσα κρίση είναι ότι βασιζόμαστε, οι αγορές βασίζονται υπερβολικά στις βαθμολογήσεις αυτές και αυτό σημαίνει ότι οι αξιολογήσεις του δημοσίου χρέους, ακόμα και από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, δεν λαμβάνονται υπόψη. Υπάρχει κίνδυνος ε, πολιτικής μεροληψίας και επιρροής, αλλά υπάρχουν και ορισμένα γεγονότα που καταγράψαμε κατά τη διάρκεια αυτής της ε, κρίσης. Αυτή η υπερβολική, ε, το ότι βασιζόμαστε μάλλον υπερβολικά σε αυτούς τους ε, οργανισμούς πιστοληπτικής ικανότητας, οδηγεί σε μεροληψίες, διότι πολλές φορές δεν υπάρχει σωστή λογοδοσία και πολλές φορές υπάρχουν, ε, ελοχεύουν μεγάλοι κίνδυνοι σε σχέση με το δημόσιο χρέος. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ε, υποβάλει το θέμα στο ελεγκτικό συνέδριο, διότι πρόκειται για έναν εξωτερικό, για έναν ανεξάρτητο οργανισμό. Επίσης, μιλήσατε για τον μηχανισμό χρηματο χρηματοπιστωτικής ε, χρήσης. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο υπάρχει και σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ συστημάτων πιστοληπτικής ικανότητας. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μόνο τις πιστοποιημένες, τους πιστοποιημένους οργανισμούς που να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικά στοιχεία έτσι ώστε να μην έχουμε βαθμολογήσεις όταν δεν ζητούνται ρητός. Αυτά είναι τα σχόλια του κυρίου Τζάνι Πιτέλα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ε, Ευχαριστούμε, Άννη. It's not present. Ashley Fox is neither present, but I will give the floor then to Kay Swinburne. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι ε, παρατηρήσει που θα σα κάνω είναι του κύριου Φόξ, ε, δεν είναι δικέ μου. Ο κύριο Φόξ ε, ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι παρόν κατά τη διάρκεια τη σημερινή συζήτηση. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δόκτωρα Κλίν για τη συνεργασία του και την πολύ χρήσιμη συνάντηση αυτή τη βδομάδα. Θέλουμε να βελτιώσουμε την λειτουργία των οργανισμών αξιολόγηση πιστολογική ικανότητα στην Ευρώπη και γι' αυτό ε, επικροτούμε τον θετικό ρόλο της ΕΣΜΑ και την ενθάρρυνση της, ε, του ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή αγορά. Πιστεύουμε ότι, ένας ότι ένα Ευρωπαϊκό Ίδρυμα ε, Αξιολόγησης Πιστολεπτικής Ικανότητας θα πετύχει τους στόχους μας και θέλουμε να τονίσουμε την ανεξαρτησία του Ιδρύματος αυτού. Επίσης, μετά από την αρχική χρηματοδότηση να μην λάβει περαιτέρω επιδότηση. Εάν ε, φανεί ανεπιτυχής ε, επιτυχές το Ίδρυμα, τότε θα πρέπει να ε, το αφήσουμε να αποτύχει και την ιδέα αυτή φαίνεται να στηρίζει και ο κύριος Κλίνης. Ευχαριστώ. Thank you very much, Miguel Ο Miguel θα επικεντρωθώ σε δύο θέματα, δύο πτυχές της πρότασης, η οποία ενέχει πολλά θετικά στοιχεία. Νομίζω όμως ότι το πραγματικό πρόβλημα είναι η έκφραση που χρησιμοποίησε ο κύριος Γκοζές όταν μίλησε για τοξικότητα. Είναι γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με πληθώρα βαθμολογήσεων το ζήτημα είναι κατά πόσο όμως θα φτάσουμε σε μία έκθεση η οποία είναι σκόπιμη σε σχέση με τις ε, βαθμολογήσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν πρωτίστως είναι το δημόσιο χρέος. Όπως είπε και ο κύριος Κλίνς, το δημόσιο χρέος για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν χρειαζόταν να βαθμολογηθεί. Και τα δημόσια χρέη οδηγούν σε άλλα ε, στοιχεία που τα διαφοροποιούν. Δηλαδή το δημόσιο ε, χρέος το καταβάλει ο φορολογούμενος. Δεν καταβάλει το κόστος ο επενδυτής, ο οποίος κερδίζει χάνει. Το δημόσιο χρέος καταβάλλεται από τον φορολογούμενο καθαρά και αυτό αποτελεί μία ιδιαιτερότητα. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν πολύ λίγα χρηματοοικονομικά προϊόντα που να έχουν μία σαφή εικόνα πληροφοριών ως προς τους ε, εμπλεκόμενους, ενεχόμενους κινδύνους σε σχέση με την έκδοση δημοσίων ομολόγων. Άρα, από πλευράς προσφοράς δεν υπάρχει ένα πρόβλημα πληροφόρησης. Κατακλείζεται ο τύπος, όμως από πλευράς ζήτησης έχουμε να κάνουμε με θεσμικούς ε, επενδυτές και με μεγάλα καρτέλ τραπεζών. Μιλάμε για ελεγχόμενες αγορές και σε αυτούς τους διαγωνισμούς δεν συμμετέχει το κοινό, αλλά τα μεγάλα καρτέλ, τα οποία πρέπει να έχουν εσωτερικές αναλύσεις, ανάληψης κινδύνου. Εάν θέλουμε να αποτοξινώσουμε ορισμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα, Αυτά τα προϊόντα είναι τα δημόσια χρέη, το δημόσιο χρέος. Γι' αυτό θα πρέπει τα 27 κράτη-μέλη να αποφασίσουν ότι δεν θα πληρώνουν, δεν θα καταβάλουν το αντίτιμο των τίτλων τους. Είναι καθαρά πολιτική απόφαση. Δεν νομίζω ειλικρινά ότι μπορούμε να απαγορεύσουμε από τους ε, επενδυτές να αγοράζουν τίτλους. Εν πάση περιπτώσει, οι κρατικοί τίτλοι είτε έχουν χαμηλό είτε υψηλό αντίτιμο έχουν συγκεκριμένες εφαρμογές. Άρα το σημείο κλειδί είναι ακριβώς αυτό. δεν μπορούμε να θεωρήσουμε το δημόσιο χρέος ως ένα δομημένο ομόλογο. Τώρα, σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, εγώ έχω ορισμένε επιφυλάξεις για αυτό το Ίδρυμα, που έγκυται στο εξή. Νομίζω ότι όλα τα Ιδρύματα Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας δεν πληρώνονται από τον εκδότη, αλλά από την αγορά. Και μόνο αν η αγορά ζητά βαθμολόγηση γίνεται. Εδώ μιλάμε για τις χρηματοοικονομικές αγορές. Ποιος ε, επενδύει, ποιος αγοράζει. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ίδια η βαθμολόγηση πολλές φορές έχει, ενέχει ένα στοιχείο τοξικότητας, διότι υπάρχουν συμφέροντα πίσω από τη βαθμολόγηση. Άρα δεν έχει νόημα να χρηματοδοτήσουμε με το δημόσιο χρήμα ένα ίδρυμα το οποίο θα είχε ιδιωτικό χαρακτήρα. Αυτό θα ήταν απαράδεκτο. Τη στιγμή που μιλάμε για ένα ίδρυμα το οποίο χρηματοδοτείται από το δημόσιο αλλά έχει ιδιωτικό χαρακτήρα, δεν μπορεί να τύχει χρηματοδότησης από το δημόσιο χρήμα, από το δημόσιο κορβανά. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι η παρέμβαση και ο παρεμβατισμός της αγοράς. Αυτά είναι τα σχόλιά μου και σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να κάνω ορισμένα σχόλια για τις ε, τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Εκτιμώ ιδιαίτερα αυτή την εργασία του εισηγητή και νομίζω ότι θα φτάσουμε σε ευρία συνένεση. Θα ήθελα απλώς να πω ως προς την σημασία της μεθοδολογίας που χρησιμοποιούμε των ε, Ιδρυμάτων Αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και ως προς το δημόσιο χρέος, νομίζω ότι θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε τη μεθοδολογία τους, να δούμε ποια είναι η κρίση τους όταν ε, προβάλλουν τέτοια ζητήματα και να δούμε κατά πόσο υπάρχει απόκληση από τις προβλέψεις διεθνών οργανισμών. Αυτό είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Δεύτερον, όσον αφορά την δημοσιοποίηση των βαθμολογήσεων. Εάν λάβουμε υπόψη τη σημασία της αγοράς, νομίζω ότι η δημοσιοποίηση θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με προσυμφωνημένα κριτήρια ως προς την διαφάνεια και τον εμπιστευτικό χαρακτήρα. Αυτά τα δύο στοιχεία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, διότι μιλάμε για ευθύνη των ε, Ιδρυμάτων Αξιολόγησης. Πολλές φορές υπάρχουν υψηλότερες απαιτήσεις, ιδιαίτερα όταν υπάρχει υψηλό ποσοστό αμέλειας. Γιατί θα πρέπει να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο αυτοί οι οργανισμοί κατά την αξιολόγηση. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ορισμένα προσυμφωνημένα κριτήρια ως προς τα πρωτόκολλα αυτά. Και ως προς το μοντέλο αυτών των οργανισμών αξιολόγησης, νομίζω ότι ως προς ε, ορισμένα δομημένα προϊόντα δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με το παρόν μοντέλο, διότι θα πρέπει αυτός που εκδίδει να, απο, να προαποφασίσει τι μοντέλο θα χρησιμοποιήσει. Εάν υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση αρμοδιοτήτων, θα πρέπει να μην υπάρχει αποκλειστική δραστηριότητα αυτών. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε και τον ρόλο των αναλυτών, οι οποίοι πολλές φορές μπορούν να δουλεύουν για αυτούς τους, οργανισμού για αυτούς τους οργανισμούς αξιολόγησης. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε λύσεις ως προς αυτές τις συμμετοχές. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που εκφράζει ένα 70% αυτών των βαθμολογήσεων. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς μπορεί να προωθηθεί μία κατανομή. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να αρκεστούμε στην παρούσα κατάσταση. Χρειάζεται ε, δημόσια παρέμβαση, η οποία και θα πρέπει να προωθηθεί άμεσα. Ο κύριος Κλίντς έχει το λόγο για να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Το ερώτημα είναι αν ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να τοποθετηθεί. Καλά, εάν όχι, ρώτησα λέει ο Πρόεδρος, αλλά φαίνεται πως ε, δεν ενδιαφέρονται. Θα ευχαριστήσω όλους και όλους τους συναδέλφους για τα επικοδομητικά του σχόλια που ενισχύουν την πεποίθησή μου ότι στους περισσότερους τομείς θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμού που νομίζω θα ικανοποιήσουν λίγο πολύ όλους. Ορισμένοι τομείς βέβαια θα παραμείνουν όπου θα ε, υπάρχει διάσταση απόψεων και αυτή θα, αντανακ, θα αντανακλά και στην ψηφοφορία το θέμα για παράδειγμα του δημόσιου οργανισμού που θα ε, χρηματοδοτείται από χρήματα του δημοσίου που προτείνει ο κ. Εγώ δεν είπα βέβαια ότι το οργανισμός που συζητούμε τώρα θα πρέπει να χρηματοδοτείται από χρήματα των φορολογουμένων. Το άφησα ανοιχτό. Θα μπορούσα μάλιστα να φανταστώ ότι το καλύτερο θα ήταν ο οργανισμός αυτός ή το ίδρυμα αυτό να χρηματοδοτηθεί από πόρους της ίδιας της ε, οικονομίας. δεν νομίζω ότι είναι σωστό να χρηματοδοτηθεί από χρήμα των φορολογουμένων, γιατί θα γίνει μάλλον αμέσως η απόπειρα να ασκηθεί ε, επιρροή, πίεση και η αντικειμενικότητα θα πάει περίπατο. Για όλε πάντως τις προτάσεις σα, ευχαριστώ, τις έχω σημειώσει. Θα προσπαθήσω να τι λάβω υπόψη μου στις τροπολογίε Αναμένω με ενδιαφέρον την ε, συζήτηση με του ε, σκιώδει στι 2 Μαρτίου. Ευχαριστώ πολύ. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 16 Μαρτίου έτσι ώστε να συζητηθεί στην Ολομέλεια τον Απρίλιο του 2011. Συμφωνείτε. Εντάξει, λύεται η συνεδρίαση.